Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο θέμα που έχουμε στη σημερινή ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση κόμη για την στρατηγική τη ενιαίας αγοράς σε συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Mm. Κάποιο πρόβλημα έχει το μικρόφωνο. Ε? Take two. Okay. Okay. Συμβαστική τροπολογία 9, το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ, η ηλεκτρονική επαλήθευση. E Έχουμε έναν ευρωβουλευτή παραπάνω από το ΕΛΚ από ό,τι θα έπρεπε. Ωραία, ευχαριστώ, διορθώθηκε το λάθος. Ε, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτη της εμπλητρία ε, ε, ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 67 ηλεκτρονική επαλήθευση. 66, την 66. Thank you. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 της έμπλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 ε, εγκρίθηκε η 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 21 της ΕΜΠΛ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 86 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται, συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Μάλλον εγκρίνεται 12 της έμπλη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, 2. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 105. Απορρίπτεται. Έμπλ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. That's passed. Second part in... Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ.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 μου είπαν ότι την 101, 102 και 103 έπρεπε να τις ψηφίσουμε. 101 λοιπόν υπέρ, κατά, 101 στην σελίδα 11. Φαίνεται ότι είναι συμβατές με την τροπολογία 100 που υπερψηφίσαμε. 101 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά α, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Την 103 ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Ζήτω συγγνώμη. Έχουμε φτάσει στη συμβαστική τροπολογία 12 στη σελίδα 14. Υπέρ. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε τώρα στην 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 καταπίπτει. Ε, συμβαστική τροπολογία 22 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ επαλήθευση. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές κατα... ε, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ, μπερδεμένα φαίνονται τα πράγματα. Παρακαλώ. 150. That has fallen. Απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 155 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά Νομίζω ότι, ότι απορρίπτεται. Η 158 καταπίπτει. 159 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 15, το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται. 170 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. όχι, απορρίπτεται, συγγνώμη, να την επαληθεύσουμε. That falls. Απορρίπτεται 173 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 κατά πίπτη 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 19 υπέρ Η 19 της Επιτροπής Απασχόλησης καταπίπτει. 33 ε, υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. E Απορρίπτεται. Έχουμε πάλι έναν ευρωβουλευτή παραπάνω από ό,τι πρέπει από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, διορθώθηκε το πρόβλημα. Καταπίπτει λοιπόν. Ε, τροπολογία 180 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 180. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 191 175, 156, 157, 158 θα πρέπει να τους ψηφίσουμε στη σελίδα 20, διότι είναι συμβατές. 155 έως 158. Η 154 εγκρίθηκε, οπότε καταπίπτουν. Είναι συμβατές όμως. με την 153. Πρόεδρος, εγκρίναμε την τροπολογία 154 και μου λένε ότι 155, 157 και 158 καταπίπτουν για το λόγο αυτό. θα παρακαλούσα τους συμβούλους σας να το ελέγξουν, διότι εφόσον εγκρίναμε την 154, ο κατάλογος ψηφοφοριών μου λέει ότι οι 155, οι 157 και οι 158 καταπίπτουν. Η 154 καταπίπτει. Όχι, λέει η Πρόεδρος, η 154 εγκρίθηκε. Θα προχωρήσουμε και ε, ας το ελέγξουν αυτό οι σύμβουλοι σου την ώρα που ψηφίζουμε πρωτού φτάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Όχι, μπορώ πολύ εύκολα να το ψηφίσω. Η 152 εγκρίθηκε. Ωραία. Η 154 καταπίπτει. Α, μάλιστα. Ζητώ συγγνώμη, έχεις απολύτω δίκιο και εγώ έχω λάθο και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Γι' αυτό πράγματι δεν έπρεπε να ψηφίσουμε την 154. Πρέπει να ψηφίσουμε την 155 υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. 155 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 158 υπέρ κατά Ζητώ συγγνώμη και την 156 πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ, 156. Η 156 καταπίπτει. Η 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνοψίζω. Στην παράγραφο 12 εγκρίθηκαν οι τροπολογίες 153, 155, 156 καταπίτη, εγκρίθηκε 157 και εγκρίθηκε 158. Και επίσης εγκρίθηκε η 159 για την παράγραφο 12α. Ζητώ συγγνώμη, είναι πολύπλοκη η κατάσταση. Νομίζω ψηφίσαμε την συμβαστική τροπολογία 16 στη σελίδα 27 ε, και προχωράμε στην 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι καταπίπτει, νομίζω ότι απορρίφεται, αλλά στο ελέγξουμε. 196 ελέγχουμε. this close. That falls. <coughs> So we're now going to um, Απορρίπτεται και προχωράμε στην 207 στη σελίδα 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 209 Όχι, πρέπει να τις ψηφίσουμε όλες αυτές. Ε, θέλετε να τις ψηφίσουμε ε, όλες μαζί την 209 ε, έως 216. Όχι. Λοιπόν, 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 ψηφοφορία κατά τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 219. Το τελευταίο κομμάτι υπέρ κατά α, αποχές εγκρίνεται. Να το επαληθεύσουμε. That Εγκρίνεται. 221. Καταπίπτει. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 228 καταπίπτει. 229, 230, 231 και 232 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19. 238 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. 238. Απορρίπτεται. 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 240 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 της Επιτροπής Αποσχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 της ε, Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 37 Εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 2.44 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 245 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 246 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 247 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 254 Καταπίπτει. 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ κατά... Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Thank Απορρίπτεται. Ζήτω συγγνώμη, μάλλον. Η 271 καταπίπτει 4 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 272 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 273 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 275 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 276 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Falls 277. 277. Απορρίπτεται 276. 277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 279 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24 ε, σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 295 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 296 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 298 και 299 καταπίπτουν και οι επόμενες καταπίπτουν όλες μέχρι που φτάνουμε στην 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 309 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 312 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 313 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. That's passed. 314. Εγκρίνεται 314 υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ και τις 314. Α, όχι, συγγνώμη, εγκρίνεται. Εγκρίνεται 3.14, 3.15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 317 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ της 317. Απορρίπτεται. 24 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά... Η 24 καταπίπτει, 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 318 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 320 πίπτη. 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 322 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 323 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 324 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 326 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε και τις επόμενες. 327 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 328 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. 329. Απορρίπτεται. 329 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 330 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Yes, it's passed. Εγκρίνεται 331 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 της Επιτροπής Αποσχόλησης υπέρ κατά... Α, καταπίπτει 31. 332 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 333 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 334 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 335 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 336 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται 337 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 338 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 341 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 342 υπέρ κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται. 25 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. 25 της Επιτροπής Απασχόλησης. Εγκρίνεται. Αλλά με πολύ μικρή διαφορά. 11 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 433 λέει η Πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 344 υπερκατά κατά αποχές απορρίπτεται, 345 υπερκατά κατά αποχές απορρίπτεται, 346 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 347 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. 348 υπέρ 348 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 349 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 350 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 351 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 354 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. That falls. Απορρίπτεται. 355 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 356 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 357 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 358 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 360 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 361 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 363 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 351 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 23 σε τρία τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Εγκρίνεται και το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 374 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ 374 Sorry, falls. Thank you. Απορρίπτεται. 376 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 375 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 378 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 379 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 380 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ένα της Επιτροπής Αποσχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά... Νομίζω ότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε την 2 της Επιτροπής Απασχόλησης. Τροπολογία 2. Τροπολογία 2. Start again. It's so... Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τροπολογία 2. Πρόκειται για αιτιολογική αναφορά 8α νέο. Υπέρ. Τρεις δεν ψήφισαν από τους παρόντες. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Νέα, κάμερα έχουμε. Άμα σφωτογραφίζετε. Λοιπόν, προσέξτε, σας φωτογραφίζουν. Σε λίγο θα έχουμε και τηλεκατευθυνόμενα ε, ε, αεροσκάφη. Εν πάση πτώση. Τροπολογία 3. Υπέρ. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Yeah, Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 και 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. C2 ε, τη Επιτροπή αποσχολή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ να ε, το επαληθεύσουμε. Την 10. Falls. Απορρίπτεται 11. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ήθελα να το ελέγξουμε και αυτό, παρακαλώ. That falls.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 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. το δεύτερο τμήμα της, της συμβαστικής 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 ε, καταπίπτει. 47 υπέρ 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α τη Επιτροπή Απασχόληση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κάποιος έχει σηκώσει την καρτέλα του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθες. Απέστειλα ένα έγγραφο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθε λοιπόν έστειλα ένα έγγραφο προ την γραμματεία. Στις γραμματείες μάλιστα ε, της και των σκιωδών και βάσει του 156.3 του κανονισμού είχα παρουσιάσει μία άποψη και μία ψηφοφορία μειονοτήτων, μειοψηφίας για να την ψηφίσουμε. Να διαβάσω λοιπόν τι προβλέπετε πρέπει να περαστεί ακόμα, μηχανισμοί όπως η ιστορική αγορά οδήγησαν ε, σε απομάκρυνση των μηχανισμών ρύθμισης της ε, αγοράς και στην ε, ασυμμετρία σε ό,τι αφορά την οικονομία οδήγησαν σε δημιουργία φορολογικών παραδείσων και απορριθμίσεις και συγκέντρωση του κεφαλαίου η οποία και προωθείται η ιστορική αγορά, δεν χρησιμοποίησε υλικό προπαγάνδας εις βάρος της αλληλεγγύης και της συνεργασίας και έτσι προωθήθηκε ξεκάθαρα ο φιλελευθερισμός. Αυτό προς εις βάρος της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας των προτύπων εργασίας, των κοινωνικών και ηθικών αξιών, οι οποίες και καταστράφησαν και η φορολογική πολιτική θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη και επειδή δεν υπάρχει ανάπτυξη, αυξήθηκε η ενεργεία, αυτό έπλεξε ιδιαίτερα στους τις χαμηλόμισθους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στρατηγικές για την ιστορική αγορά. Είμαστε κατά όμως γιατί πρόκειται για κάτι καπιταλιστικά κινήματα τα οποία θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκέντρωση του πλούτου σε μεγάλους ομίλους, σε απελευθέρωση και εκμετάλλευση στις ε, οικονομίες ε, των κρατών μελών. Και υπάρχουν λοιπόν στοιχεία τα οποία επιβάλλονται στους ε, εργαζόμενους, αλλά ουσιαστικά τα συμφέροντά τους σε καμία περίπτωση δεν προστατεύονται. One moment. Ένα λεπτό. Να σας διαβάσω τον κανόνα υπαριθμών 56. Στον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Όταν η γνώμη της Επιτροπής ε, δεν είναι ομόφωνη, η έκθεση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ε, σύνοψη και ε, της γνώμης της μειοψηφίας. Αυτές θα εκφράζονται αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία πάνω στο σύνολο του κειμένου. Κατόπιν αιτήματος ε, των ε, συντακτών μπορεί να αποτελέσει ε, αντικείμενο μιας γραπτής δήλωσης 200 λέξεων το πολύ που θα επισυνάπτεται στην δήλωση και η Πρόεδρος, εγώ δηλαδή, θα επιλύει οποιασδήποτε διαφωνίες προκύψουν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Η Γκουε στο σύνολό τη ζητάει αυτή την ε, γνωμοδότηση. Όχι, ο κανόνας αναφέρεται σε μέλος, όχι σε ε, πολιτική ομάδα. Δεν είναι γνώμη της πολιτικής ομάδας. Ναι, αλλά λέει ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σύνοψη της ε, γνώμης της μειοψηφίας. Κατόπιν αιτήματος των συντακτών της. Πρόεδρος, ναι. Αλλά Εάν θέλουμε να επισυνάψουμε τη γνώμη της μειοψηφίας, θα συμπεράνει κανείς ότι οποιοδήποτε δεν συμφώνησε στο σύνολο της έκθεσης αυτής, συμφωνεί με όλα όσα διαβάσατε. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν άλλοι ευρωβουλευτές που δεν επιθυμούν... Ένα λεπτό παρακαλώ, περιμένετε. Που επιθυμούν είτε να απόσχουν ή να καταψηφίσουν την έκθεση αυτή, που δεν συμφωνούν όμως με τη δήλωσή σας. Υπάρχει κάποιος από αυτούς που δεν θέλουν να υπερψηφίσουν την έκθεση αυτή, που δεν συμφωνούν με την δήλωση του κυρίου Ευρωβουλευτή. Με τα κόκκινα του κυρίου Πεμέντο Λόπες. Mr. Pimenta Lopez. Um Πρόεδρε, κοιτάξτε, είναι κανονική αυτή και φυσιολογική αυτή η διαδικασία. και πολλέ φορέ επαναλαμβάνονται στι επιτροπέ. Υπάρχουν απόψεις των μειοψηφιών οι οποίε πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτέ στην έκθεση. Αλλά εδώ πέρα αναφέρουμε τον υπογεγραμμένο. Δεν ε, υπάρχει θέμα του να είναι τοποθέτηση τη ε, μειοψηφία η οποία θα πρέπει να φέρει υπογραφή και άλλων. Μπορεί να υπάρχουν διάφορε τοποθετήσει ε, μειοψηφίων και ενδεχομένω να υπάρχουν διάφορε ιδεολογικέ αξιολογήσει οι οποίε είναι διαφορετικέ και από πλευρά ε, δική σα. Η πρόεδρο. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί, δεν το θεωρώ φυσιολογικό και εξ όσων καταλαβαίνω από το κείμενο, όταν μιλάμε για άποψη μειοψηφία, αυτό που εννοείται είναι ότι η άποψη τη μειοψηφία συγκεντρώνει τι απόψει όλων όσων δεν υποστηρίζουν την έκθεση. Να ακούσω και τον κύριο Αντωνέσκο και τον κύριο Σφάμπ. Ναι, κοιτάξτε, εγώ πραγματικά ενίσταμαι στι ανοησίε αυτέ. Στις ανοησίες αυτές. Η πρόεδρο. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που εκφράζετε την άποψή σα ε, αλλά θα ήθελα πραγματικά να σιγουρευτώ ότι αυτό αποτυπώνει τι απόψει όλων όσοι δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν. Κύριε Σφαπ, Βίκυ, κοιτάξτε να είμαι λίγο πιο ευγενικό από τον Τόνι, αλλά καταρχά ε, ο κανονισμό προβλέπει με ε, γραπτή δήλωση με λιγότερη από 200 ε, λέξεις. Δεν νομίζω ότι είναι δημοκρατικό να παίρνει το λόγο κανείς και να μιλάει δύο λεπτά κατά την διάρκεια της τη ψηφοφορία και η δημοκρατία έχει να κάνει με πλειοψηφίε. Δεν έχει πλειοψηφίε. Αν θέλει να μπει αυτό γραπτά στην έκθεση, α το βάλουμε. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά να δούμε πώ θα διαμορφωθεί η πλειοψηφία στο τέλο τη ψηφοφορία, γιατί μπορεί τελικά να είναι ομόφωνη η υπερψήφιση. Οπότε τι νόημα έχει που το συζητάμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάλτον. Ήθελα να πω και εγώ όπως το ίδιο όπως είπε και ο, ο Ανδρέας. Αξ' ε, λέει ο κανονισμός είναι γραπτή η δήλωση. Σας έδωσε, κυρία Πρόεδρε, γραπτή δήλωση ο συνάδελφός. Για να δούμε αν μπορούμε να ξεκινήσουμε καν. Η Πρόεδρος. Εγώ πώς ερμηνεύω το κείμενο. Ε, μάλλον απεστάλλει στους κοιόδης η γραπτή δήλωση και στη γραμματεία, προσθέτει ο κύριος Ευρωβουλευτές. Ναι, αλλά εγώ δεν το έχω δει, λέει η Πρόεδρος. Μία σαφή ερώτηση έχω να κάνω. Υπάρχει κανείς εδώ στην αίθουσα, ο οποίος σκοπεύει να μην υπερψηφίσει την έκθεση, που σκοπεύει να καταψηφίσει ή να απόσχει και που δεν συμφωνεί με τη δήλωση που μόλις ακούσαμε. Μάλιστα υπάρχει. Πολύ ωραία. Στην οποία περίπτωση πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορώ να δεχτώ την δήλωσή σας ως ε, αντιπροσωπευτική όλων των ε, ε, απόψεων της μειοψηφίας. Πρόεδρε, πρόεδρε, κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για την εφαρμογή ενός άρθρου. Λίγο αντίθετο με αυτά που λέγεται, λέγονται εδώ, γιατί θα πρέπει επιτέλους να μπει λίγη δημοκρατία εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο. Ένα τέτοιο άρθρο Άμα υπάρχει ομοφωνία στην ψηφοφορία μια έκθεση, θα πρέπει να εκπροσωπούνται και οι μειοψηφικές απόψεις στον πληθυντικό ή απόψει της μειονότητας, των μειονότητων. Δεν προβλέπετε λοιπόν τίποτα τέτοιο όπως αυτά που λέτε κατά πόσον θα καταψηφίσουν κλπ. Όχι, μιλάμε για τις απόψεις των όσων προσυπέγραψαν την ε, δήλωση η μου δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Έστειλα στη γραμματεία, στην συνεισηγητρία, στις κοιόδες συζητητές, όλοι ενημερώθηκαν. Και στη φάση της ε, ψηφοφορίας θα πρέπει να γίνει παραπομπή στο άρθρο αυτό και θα πρέπει να διαβαστεί, να ακουστεί και αυτή η άποψη, η μειονοτική. Κοιτάξτε Βίκη, ο κύριος Ντογιόγκ, είπα ήδη ότι η δήλωση δεν είναι εξ ονόματος της ομάδας ούτε με εκφράζει. Είναι προσωπική δήλωση ενός βουλευτή και θα ζητούσα εφόσον είναι δυνατόν αν το όνομα του κυρίου Λόπες το οποίο ε, αναφέρεται στην ε, δήλωση στη... αν αυτό ε, προσθεθεί αυτή στην έκθεση. Αυτό αποτελεί πρόβλημα. Κοιτάξτε, λέει η Πρόεδρο, αυτό το θέμα. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι το εξή. Αν το ονομάσουμε αυτό, αν το χαρακτηρίσουμε μειοψηφική άποψη, θα φαίνεται ότι είναι σαν σύνοψη όλων των ε, μειοψηφικών τοποθετήσεων. Και ο κανονισμός προβλέπει ότι μπορεί να υπάρχει μειοψηφική άποψη που θα εκφράζει την μειοψηφία. όπου η τοποθέτηση της, Ευρω... της Επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η έκθεση θα αποτυπώνει επίσης συνοπτικά την άποψη της μειονότητας. Τελεία. Ναι, κοιτάξτε, μιλάω αγγλικά, διαβάζω αγγλικά, το στο καταλαβαίνω. Η μειοψηφική άποψη θα εκφραστεί και μπορεί να υποβληθεί σε γραπτή δήλωση που δεν θα ξεπερνά τι 200 λέξεις ως προσάρτημα. Να κάνω μία πρόταση. Θα το συζητήσω αυτό με τη δυναμική υπηρεσία μετά την ψηφοφορία. Κατανοώ το δικαίωμα των όσων δεν υποστηρίζουν την έκθεση να καταλήξουν από κοινού σε μία ή σε περισσότερες μειοψηφικές τοποθετήσεις. Ε, δέχομαι το δικαίωμά σας, αυτό και το σέβομαι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείτε να μιλήσετε εξ ονόματος όλων όσοι δεν υποστηρίζουν την έκθεση αυτή. Θα προτείνω λοιπόν, Ντένις, όλοι όσοι δεν υποστηρίζετε την έκθεση, να συναντηθείτε εκ των υστέρων και να προτείνετε ή μία ή περισσότερες μειοψηφικές τοποθετήσεις. Αλλά θα συμβουλευτώ τη νομική υπηρεσία επ' αυτού. Αν συμφωνείτε και να περάσουμε στην ψηφοφορία, λοιπόν. Πολύ ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν στο, επί του συνόλου του κειμένου. Η κυρία Μίτση ζήτησε το λόγο. Αν σωστά κατάλαβα, λέει η κυρία Μίτση, κάποιο είπε ότι η δήλωση αυτή απεστάλλει στου κοιότε. Θα ήθελα να σα πω ότι εγώ δεν έλαβα οποιαδήποτε τέτοια δήλωση να ληφθεί υπόψη αυτό. Και επίση ε, θα επιψηφίσουμε την έκθεση και άρα δεν συμφωνούμε με τη δήλωση του Ευρωβουλευτού. Η ΕΝΕΦ δήλωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι είναι σαφές το νομικό κείμενο. Εγώ είμαι νομικός ε, και θεωρώ ότι το κείμενο αυτό δεν ε, μπορεί να γίνει αποδεκτό και θα ήθελα να μπει αυτό στα πρακτικά μάλιστα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν επί του κειμένου στο σύνολό του. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρε. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Να προτείνω ότι οι τρεις που καταψήφισαν θα πρέπει να συνειδηθούν και να αποφασίσουν κατά πόσον θέλουν να προβούν σε δήλωση ή διαφορετικές δηλώσεις για την άποψη της μειοψηφίας. Ε, ε, ε βέβαια, φαντάζομαι ότι είχαμε καταψηφίσει για το 2016 ε, αφού δεν είμαστε χώρα κομμουνιστική πάντως τέλος πάντων εγώ να ευχαριστήσω λέει κύριε Κόμη όλους μια που το θέμα αυτό ε, συγκέντρωνε την Γενική Συνένεση ε, άστα λαβίστα στα σιέμπρελ καλά προχωράμε λέει τώρα η Πρόεδρος στην έκθεση Τρεμπέσιος που αφορά τα εικονικά νομίσματα Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, παράγραφος 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ευχαριστώ. Um, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ κατά. Αποχές. Έλεγχος. Um, ε, απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική. Πέντε υπέρ κατά... Δεκαοκτώ υπέρ κατά αποχές. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 18 λέει ο Πρόεδρος. Και το 19. Can you all vote? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Καταπίπτει. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 30 30 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 31 ε, um, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος και απορρίπτεται στο 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα. Έχουμε άλλες τρεις ψηφοφορίες. Και άλλοι τρεις να ψηφίσουν. 31 υπέρ κατά θέλει Ε, θέλεις το λόγο, Αντρία. Απλώς να δώσω συγχαρητήρια ε, για την ε, έκθεση και για την έγκριση. Και επίσης νομίζω θα πρέπει να ξεχαρίσουμε ότι ε, βεβαίως και σεβόμαστε στο Κοινοβούλιο την ε, μειοψηφία. Αλλά θα πρέπει να μπορούμε να κατεβάσουμε κάποιες τροπολογίες ή δάλλως κάποια ε, δήλωση. Νομίζω ότι από πλευρά κανονισμού αυτό είναι το, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ιδίω όσον αφορά την έκθεση για την ενιαία αγορά. I do respect the minority's right to make a statement, but not on behalf of everybody who voted against the report. Επομένως, αυτό και για όλους όσους ψήφισαν κατά, οπότε θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι ε, έτσι το έχετε συμφωνήσει και, και μπάστα. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση Τσέσακ όπως είπαμε, θα πρέπει να απευθυνθούμε στην νομική υπηρεσία. ΣΕΖΑΚ. Η έκθεση για παράνομες πρακτικές στο εμπόριο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 81 υπέρ 81, 83 και 306 υπέρ κατά χες ε, νομίζω είναι οριακό το αποτέλεσμα κάνουμε έλεγχο That falls. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «308 υπέρ κατά αποχές και πάλι 308 υπέρ κατά αποχές κρίνεται». Θέλετε να κάνουμε έλεγχο. Και απορρίπτεται παρά μία ψήφο. 307 υπέρ. Υπέρ, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. και απορρίπτεται 93 υπέρ. Κατά έλεγχος για τον 93. και εγκρίνεται. 94 υπέρ. ...95 απερίφθη... ...331 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται... ...101 υπέρ κατά... Check. passed. Εγκρίνεται. 98. In favor. Υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για το 98. Εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά Έλεγχο. Okay, Α, συμπαθούμε γιατί μου είπαν ότι αυτέ. 97 ε, ε, έως 332 έχουν απορριφθεί 333 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 333 334 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 335 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 107 είναι γλωσσικού χαρακτήρα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος.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 Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 337 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Falls. Το 339 υπέρ, κατά, έλεγχος. Απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά και έλεγχος. Passed. 114. 114. Υπέρ. Sorry. Άρα, εγκρίθηκε το 116. Ωραία, εξοικονομήσαμε χρόνο. 121. 121 121 121. ε, υπέρ κατά και εγκρίνεται 121 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 344 υπέρ κατά έλεγχος That's passed. 127 in... 127. So hold on, these four down to compromise 9. In... Συμβαστική 9. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μία προσθήκη υπέρ, κατά, έλεγχος. 135. That's passed. Εγκρίνεται. 145. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Η υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 158. Okay, that's adopted εγκρίνεται. 12. Συμβαστική 12. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ε, 170. Υπέρ κατά έλεγχος για το 170. Zero. One some zero. Uh, και εγκρίνεται. In favor. Κατά. check. και απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να κάνουμε έλεγχο για το 180 και το 357. Άλλοι τρεις, άλλοι δύο να ψηφίσουν και απορρίπτονται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, συμπαθάτε με. Πρώτα να ψηφίσουμε και το 357. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182. Υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται είναι σε 182 και 183 να κάνουμε έλεγχο για τις 182 και 183 και εγκρίνονται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές και απορρίπτεται 188 υπέρ κατά έλεγχος That's Και γίνεται 189 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος 189. That falls. Απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 360 υπέρ κατά έλεγχος. Sorry, that falls. Um, compromise 15 in... Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 εγκρίνεται. 362 υπέρ ε, κατά έλεγχος. 362. Falls. Και απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Falls. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα προείπνονται όλα με το 207. Υπέρ, κατά, έλεγχος για το 207. Και εγκρίνεται. 208. Υπέρ, κατά, έλεγχος. και απορρίπτονται. Δεκαέξι συμβαστική υπερκαταποχές συγκρίνεται. Διακόσια δέκα υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος. για το 219 και απορρίπτεται. 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 225. και απορρίπτεται. 374 υπέρ κατά αποχές και απορρίπτωται αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο και απορρίπτωται 226 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 226 Απορρίπτεται. 375. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. This falls. 227. 227. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. και απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 α εγκρίνεται 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για το 240. Και απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές και απορρίπτεται 379 υπέρ κατά αποχές και απορρίπτεται έλεγχος για το 379 απορρίπτεται 380 υπέρ κατά Έλεγχος για το 380. Passed. 381 in favor. Mm. Υπέρ, κατά, για το 380 έλεγχος. 381. 381 έλεγχος. Και εγκρίνεται. 382 υπέρ, κατά. Αποχές. έλεγχος, αν και νομίζω ότι εγκρίθηκε. 382. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 386 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται Συμβαστική 19. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 269. 269. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά έλεγχος. 270. Απορρίπτεται. 392. 392. κατά. Έλεγχος. 392. Εγκρίνεται. 394 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Έλεγχος. 394 και απορρίπτεται. 395 υπέρ κατά άποχες έλεγχος πολύ μπερδεμένα τα πράγματα λέει ο πρόεδρος 395 um, και απορρίπτεται 396 υπέρ Κατά. Έλεγχος. Απορρίπτεται 397 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 398 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος. 397 έλεγχος. 398. Υπέρ. In favor. Against. Υπέρ, κατά, αποχές. απολύτω 398 και 272 έχει καταπέσει. 399. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε, εγκρίνεται το 399. 400 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 401 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 402 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε έλεγχο. Εγκρίνεται 403 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 273, 274, 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται έλεγχος 73, 74, 78 εγκρίνονται ένα συμβαστική ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 275, 280 και 281. Περκατά αποχές εγκρίνονται. 283. Έχει καταπέσει 276 και 287 υπερκατά αποχές εγκρίνονται. 277, 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 285 απορρίπτεται. Τροπολογία 2 εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές ε, 279, 282 και 280 όχι, όχι λέει ο πρόεδρος, μόνο το 279 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Και εγκρίνεται. 282 και 284 υπέρ κατά έλεγχος 282 και 284. «282-284 εγκρίνονται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 290 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. cost? Εγκρίνεται. 291 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος και για αυτήν 291 και απορρίπτεται 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά α, έλεγχος για τα 19. Τη 19 παρακαλώ ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. Ας ελέγξουμε και τη 18 ηλεκτρονικά. Τη 18. Εγκρίθηκε για αυτή. 22. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 22. απορρίπτεται. Μάλλον απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Απόχες. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας την ελέγξουμε να είμαστε σίγουροι για την 23. Παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίθηκε. 25 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Εγώ νομίζω ότι εγκρίνεται 25, λέει η πρόεδρος. Πάμε στη συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά αποχές. Κατοπίπτει. Έλεγχος. Όντω δεν εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Δεν δουλεύει η συσκευή σα. Για πηγαίνετε από δίπλα. Μήπω δουλεύει η διπλανή. Για δείτε λοιπόν πώ ε, καταφέρετε να ψηφίσετε στην επόμενη ψηφοφορία. 39. Υπέρ. Κατά. Έλεγχο για την 39. Εγκρίνεται. 41 και 2,96 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. 41 και 2,96. Καταπίπτει. 42 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ας ξαναδούμε τη 42 όμως, γιατί δεν είμαι σίγουρη. Πέρασε. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, 44 διορθώνει πρόεδρο υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Έλεγχο. Απορρίπτεται. 48 υπέρ Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 48. Απορρίπτεται. 2,97. Ε, Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 2,97. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Ω, κατάπισε. Με 46. Α, όχι, θα το ψηφίσουμε. 46 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. πενήντα, Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 50. Την πενήντα, Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. τι γίνεται με το ΕΛΚ και την 51. Έλεγχος. Λυπάμαι που είναι τόσο μεγάλη αυτή η διαδικασία. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Η 51 είχε περάσει. Πρέπει το δούσε. Και ελέγχουμε την 53. Πέρασε και αυτή, εγκρίθηκε. 60 ε, υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος λέω. Εγκρίθηκε. 57 υπέρ. Κατά. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε ομόφωνα. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά σου. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. εγκρίνεται. 2,99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άκρη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άκρη 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίν, ε, απορρίπτεται άκρη 3 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται Άκρη 4. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχο. Εγκρίθηκε. Άκρη 5. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχο. Εγκρίθηκε. Άγκρι 6. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Κρίθηκε η Άγκρι 6. Άγκρι 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 9. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές ε, έλεγχος. Άγκρι 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άκρη 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άκρη 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άκρη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άκρη 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος μάλλον. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την άκρη 19. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Άκρη 21 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για την άκρη 22. Εγκρίθηκε. Θέλετε να ανέξετε την 21. Όχι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 26. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και μέχρι τέλος και κάνουμε λοιπόν ε, την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. 34 <laughs> είναι οι ψήφοι υπέρ. Ο κύριος Σεζάκα. Nie, Vicky, may I, may I ask you how we do proceed with να ρωτήσω τι θα κάνουμε με τις επόμενες ψηφοφορίες, διότι δυστυχώς οι συνάδελφοι πρέπει να αποχωρήσουν. Θα πρέπει να ψηφίσουμε. Σας προειδοποίησα ότι μάλλον θα κρατήσουν πολλοί ψηφοφορίες σήμερα. Ωραία, πολύ γρήγορα. I need, I need beer. Ένα λεπτό, εξετάζουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ τους διαρμηνείς, λέει η Πρόεδρος, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Θα ήθελα να προχωρήσουμε με τις ψηφοφορίες. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε μέχρι να καταφτάσει ο Επίτροπος. Ε, φτάνουμε λοιπόν τώρα στην έκθεση ε, Σαρανσόβα για ε, την τροπολογία 1 υπέρ εγκρίνεται, συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ εγκρίνεται, τροπολογία 2 συμβαστική υπέρ εγκρίνεται. εγκρίνεται, 17 υπέρ απορρίπτεται, 19 να επαληθεύσουμε τη 18. Okay. It's fallen. Απορρίπτεται η 18. 19. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Close It falls 20. Απορρίπτεται 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ ε, αποσύρεται η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ απορρίπτεται, καταπίπτει μάλλον, 29 υπέρ κατά αποχές, ε, να το ελέγξουμε. Μία ψήφος ακόμα απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 το δεύτερο τμήμα Ο ε, Επίτροπος θα έχει λίγο χρόνο στο τέλος της συνεδρίασης. Ε, θα επανέλθει λοιπόν. Θα προχωρήσουμε όμως όσο γίνεται πιο γρήγορα. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει. 33 ε, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34, ψηφοφορία κατά τμήματα, το πρώτο μέρος υπέρ κατά εγκρίνεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Okay. That's passed. And the second part. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία... Συμβαστική τροπολογία 7, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50, υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Pass.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 Καταπίπτει. Συμβαστική 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67, yes, we'll check 67. ηλεκτρονική επαλήθευση της 67. Εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 κατά πίπτη. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 καταπίπτει λέει η Πρόεδρος, 94 υπέρ κατά 95 υπέρ κατά η 94 εγκρίθηκε 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95, συγγνώμη, απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το σύνολο της ε, γνωμοδότησης ψηφίζουμε τώρα. How many of these Έκθεση Dalton. Ε, συμβαστική τροπολογία 3. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος, δεν ακούμε. Βλέπετε τα αποτελέσματα της έκθεσης Σαρανσόβα. 30 ψήφισαν υπέρ, 5 ψήφισαν κατά. Ο επίτροπο βρίσκεται έξω από την αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε την έκθεση, της, ε, την έκθεση Dalton. Θα πρέπει όμω να προχωρήσουμε γρήγορα. Ωραία, προχωράμε. Συμβαστική τροπολογία 3, υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4, υπέρ. Εγκρίνεται. 36, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 4 εγκρίθηκε. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 52 καταπίπτει, 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 55 υπέρ 55 η 55 δεν καταπίπτει. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58, 59 έχουν αποσυρθεί. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 καταπίπτει. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 71. Απορρίπτεται. Σας ευχαριστώ. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά εγκρίνεται 86 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 11 εγκρίνεται 91 ε, κατα, απορρίπτεται συμβαστική 12 ε, εγκρίνεται η συμβαστική 12 98 εγκρίνεται 13 εγκρίνεται 14 εγκρίνεται. 105 απορρίπτεται. 15 συμβαστική εγκρίνεται. Συμβαστική 16 εγκρίνεται. 117 απορρίπτεται. 17 εγκρίνεται. 123 απορρίπτεται. 124 Απορρίπτεται. 125. 131. 131. Ε, υπέρ κατά απορρίπτεται. 132. Απορρίπτεται. 118. Όχι, συγγνώμη, συμβιβαστική 18 διορθώνει η Πρόεδρος, εγκρίνεται. 136, εγκρίνεται. 19, εγκρίνεται. 139, υπέρ της 139, παρακαλώ, κατά, ε, να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Passed. Εγκρίνεται. 140. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Εγκρίνεται. 153. Εγκρίνεται. 154. Εγκρίνεται. 155. 155. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 22 εγκρίνεται. 150 λέει η Πρόεδρε. Όχι, συγγνώμη, διορθώνει 160 υπέρ κατά εγκρίνεται. 161 αποσύρεται. 162 εγκρίνεται. 163 ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 23 εγκρίνεται. 173. Εγκρίνεται. 174. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. False. Sorry. Απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη. 175 και 76 απορρίπτονται. 178 απορρίπτεται. 177 απορρίπτεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. 177. 177. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 181 υπέρ έχει αποσυρθεί. 182 υπέρ κατά εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά εγκρίνεται. 184 όχι. 185 υπέρ κατά εγκρίνεται. 24 συμβαστική 24 εγκρίνεται. 189 υπέρ. 189. Αποσύρθηκε αρκετά αργά. Συμβαστική 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. 26 εγκρίνεται. 194 υπέρ εγκρίνεται. Η συμβαστική 27 υπέρ εγκρίνεται. 197 υπέρ εγκρίνεται. Αποσύρθηκε. 198 υπέρ εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. 199. Απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 28. Εγκρίνεται 202. Εγκρίνεται 205. Εγκρίνεται 206. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Εγκρίνεται. 1. Εγκρίνεται. 2 απορρίπτεται, 3 εγκρίνεται, 4 καταπίπτει, 6 εγκρίνεται, συμβαστική 1 εγκρίνεται, 11 εγκρίνεται, 12 και 13 καταπίπτουν, ε, απορρίπτονται 14 η ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται 15. Απορρίπτεται 16. Εγκρίνεται 17. Εγκρίνεται 18. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Εγκρίνεται. 22. Ε, καταπίπτει 24. Εγκρίνεται 25. Καταπίπτει 26. 27 εγκρίνεται, 26 εγκρίθηκε, 27 εγκρίθηκε, 28 εγκρίνεται, 29 εγκρίνεται. Και το ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης. Ένα λεπτό ακόμα παρακαλώ. Εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και έχουμε μία μοναδική ψηφοφορία στο τελευταίο θέμα, δική μου και του κυρίου Ζουβά, για τον κοινό τελωνιακό κώδικα. Ευχαριστώ Φιλίππε, εξαιρετική δουλειά, μία ψήφος. Νομίζω ότι μόλις σώσαμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ όλους σας. How late we? Με ρώτησε λοιπόν ο επίτροπο τι συζητούσαμε και τι ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε την αναθεώρηση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τη συνολική στρατηγική για την ενιαία αγορά. Επίσης την έκταση για τις μη δασμολογικούς, μη ε, φραγμούς και για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Τα σημαντικά λοιπόν αυτά τα θέματα, όπως και η έκθεση για τα επόμενα βήματα για την εμπορική ε, πολιτική και για τα εικονικά νομίσματα ψηφίσαμε. Και η ομάδα του Επιτρόπου Μοσκοβισή έχει καταρτήσει ένα κώδικα τελωνιακό για τις μεταβατικές ε, τέτοιες ε, φάσεις για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Ήταν λοιπόν μεγάλη Μεγάλε οι σημερινέ ψηφοφορίε. Σα παρακαλώ λοιπόν, συνάδελφοι, καθίστε. Start. Um, so the, uh, next item on... Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο ε, κύριο Άνσιπ, αρμόδιο για θέματα ενίας ψηφιακής αγοράς. Τμήμα του ετήσιου διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα εργασία τη. Θα του δώσω λοιπόν παρά αυτά το λόγο, ο οποίο θα μα κάνει μια παρουσίαση και επίση ε, θα αρχίσουμε να σημειώνουμε και ποιο θέλει να πάρει το λόγο για να σα βάλουμε στον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κύριο Άντσιπ που με καλέσατε. δεύτερη συνάντησή μου είναι σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Και βλέπω ότι κάποια, κάποιοι βουλευτέ συμμετείχαν και στην πρώτη συνάντηση και τώρα λοιπόν σα ξανασυναντώ σε άλλη συνεδρίαση σε ό,τι αφορά την ενιαία ψηφιακή αγορά και το που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις προτάσεις αυτές. Θα θυμάστε όλοι ότι ξεκινήσαμε την ε, πολιτική, τη στρατηγική αυτή για την ενιαία ψηφιακή αγορά το Μάιο πέρσι και το Δεκέμβριο υποβάλαμε δύο τέτοιες προτάσεις βάσει της στρατηγικής αυτής. Και οι δύο λοιπόν αυτές προτάσεις ε, υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο και συνδέονται με θέματα αρμοδιότητος της Επιτροπής σας. Μία πρόταση ήταν για τους ε, κανόνες επικοινωνίας. Όπως ξέρετε, σήμερα έχουμε 28 πακέτα ε, κανόνων σε ό,τι αφορά την πωλήση τέτοιων αγαθών και ενδεχομένω να υπάρχουν και 28 άλλα πλαίσια για το ψηφιακό περιεχόμενο και τις σχετικές πωλήσεις. Και θα έχουμε δύο κανόνες, αφορά, δύο πλαίσια σε ό,τι αφορά τα απτά αγαθά και σε δύο σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά αγαθά. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την φορητότητα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει μεταρρύθμιση του δικαίου για τα δικαιώματα του δημιουργού. Φυσικά, οι διατάξει για τη φορητότητα δεν πρόκειται να επιλύσουν όλα μα τα προβλήματα, αλλά θα μα βοηθήσουν σημαντικά. Σήμερα 35% των Ευρωπαίων ξοδεύουν 10 ημέρες το χρόνο τουλάχιστον σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά από αυτά τα άτομα που ταξιδεύουν ε, σε άλλα κράτη-μέλη θα θέλουν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο το οποίο έχουν πληρώσει και αγοράσει. Αλλά επειδή υπάρχουν προστασία του copyright, πολλές φορές αυτό δεν γίνεται. Δεν έχουν πρόσβαση και ξέρουμε ότι 20% των Ευρωπαίων χρησιμοποιούν το VPN για να χρησιμοποιήσουν αυτό το περιεχόμενο, αλλά και το VPN δεν είναι δωρεάν. 6, 7, 8, 10 ευρώ το μήνα, 20 ευρώ το τρίμηνο πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής. Και όταν ο κόσμος ε, ε, πληρώνει το VPN δεν θεωρεί ότι κάνει κάτι λάθος, αλλά τελικά ο δημιουργός δεν αποζημιώνεται δεν ε, κερδίζει τίποτε. Και δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί εξακολουθούν να υφίστανται αυτοί οι προορισμοί τη φορητότητα. Αν ο κόσμο έχει πληρώσει μία φορά για την πρόσβασή του στο ψηφιακό περιεχόμενο στη χώρα από την οποία προέρχεται, πώ μπορεί κάποιο να έλθει και να πει ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει να έχει πρόσβαση στην ίδια μουσική, στα ίδια παιχνίδια, αθλητικό περιεχόμενο από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω όμως ότι σε κάποια κράτη-μέλη η πολιτική θα ήθελε να θέσουν κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χρονικά όρια, 7 ημέρες ή 30 ημέρες, σε πάση περιπτώσει. κατά τις οποίες θα υπάρχει αυτή η φορητότητα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστή ως ιδέα. Γιατί τα συγκεκριμένα χρονικά όρια τι θα σημαίναν για τα άτομα που ζουν στην Κοπενχάγη, στο Μάλμε, στη Σουηδία και την Δανία. Κάθε μέρα 5.000 άτομα διασχίζουν τη γέφυρα γιατί ζουν σε μια χώρα αλλά δουλεύουν σε μια άλλη χώρα. Το ίδιο μεταξύ Γαλλίας και Λουξεμβούργου. Μπρατισλάβας και Βιέννης. Κάθε μέρα ο κόσμος διασχίζει σύνορα γιατί μπορεί να δουλεύει σε μία χώρα ενώ να δουλεύει σε άλλη. Άρα, τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα αρχίσουμε να αρμονίζουμε το ποσοστό των διακοπών, Τι σημαίνει διακοπών στην Ευρώπη. Αλλά ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί το, τις κινητές του συσκευέ μόνο όταν πάει διακοπές, γιατί ορισμένοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς. Είναι σήμερα στο Βέλγιο, αύριο στην Γαλλία και μεθαύριο στη Γερμανία. Είναι αναγκαστικό δηλαδή να θέσουμε όρια για το πόσε ημέρε μπορεί να δουλεύει κανεί σε άλλο κράτο μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ένα χρόνο. Η πρόταση λοιπόν αυτή για να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χρονικά όρια, κάποιο αριθμό ημερών, ε, παραβιάζει ουσιαστικά τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί μετά θα πρέπει να αρχίσουμε να παρακολουθούμε τον κόσμο, να παρακολουθούμε το περιεχόμενο το οποίο, στο οποίο έχει πρόσβαση. Α, ακούσατε ένα τραγούδι. Ένα λεπτό 42 δευτερόλεπτα. Κι άλλο ένα. Γιατί αυτό το τραγούδι, για αυτή, αυτή η ταινία και το εξής. Θεωρώ ότι είναι ακριβή αυτή ω λύση και θεωρώ ότι αντίκειται και σε κάποιε αρχέ των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να θέσουμε λοιπόν μία σαφή διαχωριστική γραμμή η συνδρομή και ο κόσμος ε, πόσο χρόνο ε, ξοδεύει σε άλλη χώρα δεν έχει σημασία τόσο. Κάποιοι ε, το συγκρίνουν αυτό με το τέλος περιαγωγής. Εκεί θέσαμε κάποια όρια, αλλά εδώ μιλάμε για τέλος περιαγωγής, επειδή χρησιμοποιούμε το δίκτυο κάποιου άλλου. Αλλά όταν μιλάμε για υπηρεσίε φορετότητα, το, το περιεχόμενο αυτό είναι δικό σου. Το έχει πληρώσει για να έχει συνδρομή και πρόσβαση σε αυτό. Πώ μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι έχει πρόσβαση σε κάτι διαφορετικό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα πρέπει να σας πω ότι σε επίπεδο εμπρεγνωμών γνωρίζω ότι πάρα πολλές χώρες εκφράζουν ανησυχίες και αμφιβολίες σε ό,τι αφορά τον ορισμό χρονικού ορίου για τη φορητότητα. Σε κάποιες χώρες τώρα, οι πολιτικοί θα ήθελαν να ζητήσουν μεγαλύτερη περίοδο, μεταβατική περίοδο. Τώρα λοιπόν προβλέπετε έξι μήνες. Έξι μήνες θεωρώ ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι από, την 15, Ιουνίου του 2015 ε, καταρχήσαμε το τέλος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ο κόσμο ε, σταματήσει να πληρώνει τα υψηλά τέλη περιεγωγής θα θέλει να χρησιμοποιεί τι κινητέ του συσκευέ πολύ πιο πολύ σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει νομική πρόσβαση, νόμιμη πρόσβαση για αυτά τα άτομα τα οποία από 25 Ιουνίου 2017 ε, θα έχουν, δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν τέλη περιεγωγής. άλλο θα τους πρόξουμε στο να χρησιμοποιούν πιο πολύ VPN, γιατί όπως ξέρετε 68% των ε, πολιτών στην Ένωση που βλέπουν ταινίε online χρησιμοποιούν δωρεάν ε, παράνομες ε, οδούς για να κατεβάζουν τις ταινίε αυτές. Άμα χρησιμοποιούν λοιπόν πιο πολύ αυτές τις δωρεάν μορφές ε, κατεβάσματος ταινιών, ουσιαστικά δεν θα αποζημιώνεται ο εκάστοτε δημιουργός. Αυτό δεν είναι ο στόχος μας. Αυτό σε ό,τι αφορά την πρότασή μα για την φορετότητα και θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι σα ζητούμε να υποστηρίξετε το πακέτο αυτό, την πρόταση αυτή, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει μεγάλες συνέπειες. Το Φεβρουάριο του 2016 κάναμε την ε, πρότασή μας για τα 7 MHz. Αυτό συνδέεται με θέματα καταναλωτή. Σήμερα δεν υπάρχει σαφήνεια, δεν υπάρχει προβλεψιμότητα οι εμπλεκόμενοι φορείς, είτε μιλάμε για υπηρεσίες παροχής τηλεπικοινωνιών, δεν ξέρουν για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συχνότητες αυτές. Θα πρέπει να τους δώσουμε μια αλφα βεβαιότητα, μια αλφα προβλεψιμότητα. Και από το στιγμή που θα υπάρχει σαφήνεια, θα προβούν ε, και αυτοί στις επενδύσεις του. Πριν από δύο ημέρες μόλις, ξεκίνησε το πακέτο α, ψηφιακής διάστασης της βιομηχανίας. Ενδεχομένω να μην συνδέεται αυτό άμεσα με τον καταναλωτή, λένε πολλοί. Αλλά η βιομηχανία χωρί τον καταναλωτή τι είναι. Ανοησίε. Θεωρώ ότι υπάρχει λοιπόν έντονη και μεγάλη διασύνδεση. Και αυτή λοιπόν αυτό το πακέτο για την ε, ψηφιακή διάσταση της βιομηχανίας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αφορά τον πολίτη μας λοιπόν το πακέτο αυτό. Τον Μάιο ελπίζουμε στις 25 Μαΐου να παρουσιάσουμε το πακέτο μας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce. Και αυτό θα αφορά την Επιτροπή ΕΜΚΟ και πάλι. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, λάβαμε στοιχεία από τις δημόσιες διαβουλεύσεις, από έρευνες τομεακές και έγινε και μία έρευνα σε ό,τι αφορά τις αγοραπολισίες mystery shopping survey. Από αυτές τις ε, πληροφορίες προκύπτει ότι μόνο ένα τέτοιο των ατόμων που προσπαθούν να αγοράσουν υπηρεσίες για αγαθά από άλλο κράτος μέλος το πέτυχαν. Μόνο 2% των όσων απόπειράθηκαν να αγοράσουν κάτι από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν δεν είχαν πρόσβαση στα στις ιστοσελίδες αυτές. 27% των όσων είχαν πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές δεν μπόρεσαν να κάνουν την καταχώρηση τους. Γιατί δεν ήταν από τη σωστή χώρα. Δεν είχαν σωστή διεύθυνση IP. 32% των ατόμων αυτών που είχαν την τύχη να καταφέρουν να κάνουν την καταχώρησή του είχαν προβλήματα στι πληρωμέ. Δεν έγιναν αποδεκτέ οι ψηφιακές του κάρτες. Όπως ξέρετε, έχουμε το σύστημα ΣΕΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ενιαία Ευρωπαϊκό Χώρο για τι πληρωμέ. Αυτό θεωρητικά θα σήμαινε ότι δεν χρειάζεται να δεχόμαστε τέτοιε δικαιολογίε ότι α, έχουμε δυσκολίε να αποδεχτούμε την πιστοτική σα κάρτα ή οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά σε πραγματικού όρου 32% των ατόμων που κατάφεραν να καταχωριστούν τελικά δεν μπορούσαν να κάνουν πληρωμή. Δεν λέμε ότι όλοι θα πρέπει να αποδέχονται και τις ε, Mastercard και τις κάρτες Visa. Αλλά αν, μπορεί, αν αποδέχεται κανεί Mastercard Βελγίου, θα πρέπει να αποδέχεται Mastercard Γαλλία. Αλλά σήμερα αυτό αποτελεί μια σημαντική δικαιολογία για την άρνηση παροχή υπηρεσιών. Και φυσικά πολλά άτομα έχουν προβλήματα. 32% είχαν προβλήματα παράδοση 36% είχαν προβλήματα στις ε, πληρωμές. Και τελικά μόνο ένα 36,6% κατάφερε να αγοράσει κάτι από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτώ λοιπόν. Όντω μιλάμε για ενιαία αγορά, όταν τελικά ένα τρίτο μόνο του κόσμου που θέλει να αγοράσει κάτι online το καταφέρνει από άλλη χώρα. Ελπίζω να μπορέσατε να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το πολύ καλό βίντεο κλιπ που... του Μπίλκ. Βάλτε στο YouTube Μπίλκ και για αποκλεισμό. Και νομίζω ότι θα δείτε μια πολύ συνοπτική εικόνα που παρουσιάζει πολύ καλά το που βρισκόμαστε τώρα. Θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Θα θέλαμε την, να επιβάλλουμε την υποχρέωση στους παρόχους να αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό ή μεταπό. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να παραδίδει κανεί οπουδήποτε, γιατί κάποιοι είπαν ότι ενδεχομένω οι μικρομεσαίε να απαλλαχθούν από την υποχρέωση αυτή, οι μεγάλοι όμιλοι να πρέπει να παραδίδουν παντού και κάποιοι πολιτικοί είπαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε ζημία κάποιες εταιρείε. Αλλά α υποθέσουμε ότι κάποιοι λιανοπολιτέ έχουν σύστημα online πωλήσεων και παράδοσης. Αυτό θα παραμείνει ως έχει σε άλλα σημεία. Έχουν το σύστημα πωλήσεων online, αλλά δεν έχουν σύστημα παράδοσης. Αλλά έχουν κάποια υπηρεσία που παρέχει την παράδοση. Και αυτό θα παραμείνει όσο έχει. Αλλά η διακριτική μεταχείριση βάσει εθνικότητα ή βάσει χώρα έκδοση τη ψηφιακής κάρτα δεν είναι αποδεκτή. Ενδεχομένω, μια άλλη εταιρεία να μπορεί να α, πάει να πάρει τα αγαθά και να τα παραδώσει. Αν θέλω εγώ να κάνω ένα δώρο στι κόρε μου, για παράδειγμα, σήμερα πολύ απλά μου λένε ότι δεν αποδεχόμαστε την πιστοτική σας κάρτα γιατί δεν είναι εκδοθεί σα στην ε, χώρα που πρέπει. Ενώ θα υπήρχε υπηρεσία παράδοση των ε, δώρων αυτών. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μια λύση και να ξαναδημιουργήσουμε την ε, ενιαία αγορά. Πριν από 20 χρόνια το κάναμε αυτό σε πραγματικούς όρους. Αλλά τώρα η οικονομία μας και η ζωή μας ψηφιοποιείται όλο και πιο πολύ και βλέπουμε πω επανέρχονται τα σύνορα, τα εμπόδια κάθε μέρα. Θα πρέπει λοιπόν να ρίξουμε τους φραγμούς αυτούς και να δημιουργήσουμε πραγματικά ψηφιακή αγορά στην ε, Ευρώπη. Έχουμε και τη δέσμη για το ε, ηλεκτρονικό μπόρο και έχουμε το γνωτή της παράδοσης, οπότε θα πρέπει εδώ να δούμε τι γίνεται με τα βέματα αυτά τα οποία παραδίδονται. Και όπω γνωρίζετε, το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χαμηλότερε τιμέ είναι όταν μιλάμε για 2 κιλά και διασυνοριακή παράδοση είναι στις κάτω χώρες. 10 ευρώ και 50 cents. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τιμές εσωτερικού και διασυνοριακής ε, παράδοσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, στο εσωτερικό επίσης ε, υπάρχει το ρεκόρ της ελάχιστης τιμής πάλι στις κάτω χώρες αλλά υπάρχει ένα άλλο κράτος μέρος που υπάρχει διαφορά μεταξύ διασυνοριακής τιμής και εσωτερικό. 22 φορές, 22 φορές παραπάνω. Ποιος είναι σε θέση να πληρώσει τόσο ακριβά. Δεν θέλουμε να αρχίσουμε να νομοθετούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για αυτά τα θέματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, ούτως ώστε να έχουμε κάποιο είδους συγκριτικό website και να μπορούμε να ψάξουμε για 5-6 χώρες. Βέβαια υπάρχουν και 500 διαφορετικές τιμές, αλλά να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Και αυτό θα δημιουργήσει αυθεντικό ανταγωνισμό. Οπότε είμαι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές, αλλά ε, μιλάμε για 50% επιχειρήσεων και των πελατών θεωρούν ότι ο βασικός φραγμός όσο προς την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αυτές οι υψηλές τιμές της ταχυδρόμησης των ε, δεμάτων. Άρα και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Ε, Content uh, uh, uh, Δεύτερο τώρα πακέτο για τον Σεπτέμβριο. Θα είναι για το copyright η μεταρρύθμιση, οπότε εδώ θα πρέπει να είναι πιο εύκολη και συνεργειακή πρόσβαση από ό,τι είναι σήμερα. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να δούμε τη γίνεται με τις ε, παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις, τις εκπαιδευτικές, Φερρυπίν, τις ε, βιβλιοθήκες, τους ανάπηρους. Να δούμε πώς θα κυρώσουμε τη συνθήκη του Μαρακές. Μα είναι δυνατόν να μην το έχουμε κάνει αυτό. Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που την υπογράψαμε. Και τώρα υπάρχουν προστριβές ε, της θεσμικών οργάνων, οπότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να κρίνει. Δηλαδή, ποιος έχει κυρώσει αυτή τη συνθήκη στην Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Μπορεί να μην έχουμε απόφαση του δικαστηρίου ούτε το Σεπτέμβριο. Αλλά θέλουμε να περάσει αυτή η δεσμή μέτρων για να βρεθεί μια λύση. και έτσι να υπάρχει de facto εφαρμογή της συνθήκης. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Αλλά σας είπα, είναι τρομερό το ότι μια τριετία δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Άρα, μετά, ελεύθερη ροή δεδομένων. Η πρόταση διατυπώθηκε το Νοέμβριο, πολύ σημαντική ανεμπόδιση ροή των δεδομένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να παρασχεθούν ποιοτικές υπηρεσίες. Όταν έχουμε τα διασυνδεδεμένα φορτηγά, η, η Σκάνια δεν το έχει κάνει αυτό με 200.000 φορτηγά, οπότε ε, ε, κάθε δύο λεπτά υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων. Και η Σκάνια έτσι συμβουλεύει για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ε, η τεχνική κατάσταση της καμπίνας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Επίσης θα διασυνδεθούν κάποια τρένα που μεταφέρουν φορτηγά. Το θέμα είναι βέβαια γιατί θα γίνει όταν ε, διασχίζουν σύνορα αυτά τα διασυνδεδεμένα φορτηγά. Οπότε υπάρχουν πλέον οι, υπάρχει ροή των δεμένων που πια εντοπίζεται εκεί. Και στην Ιστονία, την ε, πατρίδα μου, όταν ε, περνάνε και τα φορτηγά, τι γίνεται, δεν μπορεί κανείς να έχει τα ογκώδη δεδομένα και υπάρχει και μεγάλο κόστος και για την ιατρική επίσης. Μια διάγνωση. Έχουμε ίσως τέσσερις περιπτώσεις ε, ετησίως και θα πρέπει να μπορεί ο κόσμος να συσχετίσει τα ε, στοιχεία. Θα πρέπει να πάει στα ογκώδη δεδομένα και να δει τι παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Μιλάμε Πέντε, πέντε περιπτώσεις ε, ετησίως που αυτό καθίσταται αδύνατο. Άρα χρειάζεται να δούμε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο περιβάλλον να έχουμε ελεύθερη ανεμπόδιστη ροή των δεδομένων για όλη την Ευρώπη. Αυτό να είναι εφικτό. Αλλά ακόμη περισσότερο θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον που να επιτρέπει αυτήν την ροή δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ γιατί ψηφιακό πρέπει να πει παγκόσμιο και όλοι θα ωφεληθούν από αυτή την ελεύθερη ροή των ογκωδών δεδομένων. Για τον ΦΠΑ και τη σχετική οδηγία, πειρατεία, η ανείχνευση των χρημάτων, η προέντωση εγκλήματος, όπως έχουμε την κυβερνοασφάλεια, το PPP, τη σχετική ανακοίνωση, αναθεώρηση ε, της οδηγίας για οπτικοακουστικά, μετάρρυθμιση των τηλεπικοινωνιών των σχετικών διατάξεων, σημαντικό για τους καταναλωτές. Αν θεώρησαν για τους παρόχους Αυτά για φέτος. Και διαπιστώνω με μεγάλη μου χαρά ότι πια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει κάποιες σχετικές εκθέσεις. Και θα έχουμε από τα αποτελέσματα πριν τις θερινές διακοπές. Σας ευχαριστώ και περιμένω τις ερωτήσεις σας να τις απαντήσω. Εξαιρετικά. Λοιπόν, στον ε, κατάλογο έχω διάφορους ομιλητές. Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στους συντονιστές. Ανδρέας, ε, ήθελες να πάρεις το λόγο. Εύελιν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα ζητήσει το λόγο διότι Συνήθως παίρνουν πρώτα το λόγο οι συντονιστές, αλλά να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις πληροφορίες ε, που μας έδωσε. Ε, ήταν πολύ ευρύ το φάσμα των θεμάτων που θίξατε. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρατε. Πώς θα προχωρήσουμε όσον αφορά την συμμετοχή οικονομία και τις πλατφόρμες. Τι χρονοδιάγραμμα έχουμε εδώ, διότι είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους πολίτες και φυσικά και εμάς και τους ευρωβουλευτές. Επίσης, ε, τα τρία θέματα στα οποία αναφερθήκατε, το, το επιγραμμικό περιεχόμενο, ε, τα αγαθά και η κινητικότητα είναι σημαντικά θέματα για τα οποία θα έχει διαβουλεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ως εισηγήτρια για το επιγραμμικό περιεχόμενο δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα έχουμε ολοκληρώσει πριν το καλοκαίρι, διότι είναι πολύπλοκο το θέμα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή Γιούρη και θέλουμε να κάνουμε καλή δουλειά. Εάν βιαστούμε, τελικά το αποτέλεσμα δεν ε, θα είναι βιώσιμο και δεν θα προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ελπίζω πάντως ε, να ολοκληρώσουμε φέτος. Σας ε, το λέω ενημερωτικά, πάντως όχι πριν ε, τις ε, διακοπές του καλοκαιριού. Δεν θα προλάβουμε την Ολομέλεια του Ιουλίου, για παράδειγμα. Τίθενται διάφορα ερωτήματα όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στο επιγραμμικό περιεχόμενο και τα αυτά αγαθά. Υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες, υπάρχει αρκετή ανασφάλεια όσον αφορά τους ορισμούς. Πώς ε, θα αποφασιστεί ποια θέματα ανήκουν στο ένα θέμα και ποια στο άλλο. Ε, διότι θέλουμε να αποφύγουμε την ε, νομική αβεβαιότητα και και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το DSM. Διαπιστώσαμε ότι εφαρμόζεται διαφορετικό δίκαιο ανάλογα με το αν έχει αγοράσει κανείς επιγραμμικά τα αγαθά ή όχι. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σημαντική πρόκληση το θέμα αυτό και το Κοινοβούλιο δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μπορεί να μην είναι σημαντικό θέμα για αυτούς που πολλούν μόνο ε, επιγραμμικά, αλλά για αυτούς που ε, πολλούν και επιγραμμικά και ε, αλλού, είναι αρκετή δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ πώς θα προχωρήσουμε στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Καταρχάς, όσον αφορά ε, την ε, το να μπορούν ε, να μεταφέρονται τα ε, Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, και συνήθω η ομάδα μου δεν στηρίζει τόσο πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι έχετε την σωστή προσέγγιση που προστατεύει την εδαφικότητα και επίσης αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Για μένα το βασικό πρόβλημα ωστόσο είναι ότι ε, ανησυχώ μήπως κινούμεθα προς ε, πανευρωπαϊκές άδειες. Ε, θα πρέπει λοιπόν η αδειοδότηση να γίνει σωστά. Ε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ε, δεν θα πρέπει να έχουμε χρονικά όρια, διότι έτσι ε, ε, έρεται ουσιαστικά η αιτιολόγηση της ε, πρότασης περιφορητότητας και εάν δεν καταφέρουμε να κάνουμε σωστά το θέμα του authentication, τότε δεν, ε, τότε θα αποτύχουμε. Πάντως στηρίζω την προσέγγιση σας όσον αφορά τις ε, ψηφιακέ συμβάσει Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή τη στιγμή όπου θα έχουμε διαφορετικούς κανόνες για τι πωλήσει στο διαδίκτυο ε, και εκτός διαδικτύου και υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε σε μεγάλη σύγχυση διότι βλέπουμε αρκετή ανάμειξη των, μεταξύ αυτών των δύο τρόπων πώληση. Ε, δεν μπορούμε να αναγκάσουμε επιχειρήσεις να πολλούν σε αγορές όπου δεν θέλουν να πουλήσουν και ιδιαίτερα ε, επειδή θα πρέπει να προσαρμοστούν σε κανόνες περί ΦΠΑ ε, που μπορεί να είναι πολύπλοκοι. Επιμένω όμως ότι θα πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά διότι αλλιώς θα αποτύχουμε. Επίσης όσον αφορά το να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα ως νόμισμα, διότι ε, έτσι θα καταστρέψουμε ε, το ε, μοντέλο για τα δωρεάν apps και για τις δωρεάν εφαρμογές. Επίσης, αναφερθήκατε στο YouTube, κάτι πολύ καλό, αλλά ελπίζω να μην θέλετε να πληρώνουμε για να παρακολουθούμε το βίντεο που αναφέρατε. Χθε ήταν εδώ ο επίτροπο Σότιγκερ και τον ρώτησα σχετικά με τις ε, πιθανές προτάσεις για τέλη για κάποιες ε, ε, συνδρομητικές υπηρεσίες ή το YouTube ή επίσης κάποιο φόρο για ιστοσελίδες ειδήσεων. Υποστήριξε ότι η μεγάλοι ε, εκδότες ε, αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, ε, αλλά ο λόγος μάλλον είναι ότι δεν έχουν προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Ε, Πάντω, σα παρακαλώ, μην σκοτώσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί πολλοί κόσμο στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να δεσμευτείτε ότι δεν θα επιλέξετε τη δική μα οδό, αλλά υποθέτω ότι κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο και επίσης όσον αφορά την ε, ε, ε, συμμετοχή οικονομία, σας παρακαλώ σκεφτείτε τους καταναλωτές. Έχουμε εκατομμύρια επιχειρηματίες που δημιουργούν επιχειρήσεις σε τομείς όπου πολλοί κόσμος δεν ήξερε καν ότι υπάρχουν αγορές. Σας παρακαλώ λοιπόν μην σκοτώσετε αυτή την οικονομία. Θα πάω στην τολέτα ένα λεπτό, αλλά θα επανέλθω για να ακούσω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Δυστυχώς, ε, λόγω του ότι καθυστέρησαν οι ψηφοφορίες, ε, δεν είναι πολύ παρόντες ε, εδώ κατά τη συζήτηση. Είναι όμως πολύ σημαντικά τα θέματα σας για την Επιτροπή μας και ίσως θα πρέπει να συναντιόμαστε πιο συχνά. Επίσης ε, χαίρομαι που χάρη σε εσά έχουμε ξεφύγει από τα λόγια και έχουμε προχωρήσει σε δράσεις. Βλέπουμε ήδη κάποιες πρώτες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τουλάχιστον εκ μέρους της δικής μας πολιτικής ομάδας μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προωθήσουμε τα θέματα αυτά διότι θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες μας. Αναφέρατε πολλές προτάσεις, ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα όμως ε, να γνωρίζω τις ε, απόψεις σας σχετικά με την πρόσφατη πρόταση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα πρότυπα για τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών. <clears throat> Θέλουμε να εξαλείψουμε τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Ε, κάτι τέτοιο όμως θα είναι δαπανηρό και είπατε ότι δεν προβλέπετε να υπάρξει χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι βασίζεστε σε ε, ιδιωτικές συμπράξεις και την ε, συμβολή των κρατών μελών. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν λαμβάνετε υπόψη σας και την οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη. Έχετε κάποια δεδομένα, έχετε κάποια δέσμευση από τα κράτη-μέλη στο σημαντικό αυτό τομέα. Θα ακούσουμε την Τζούλια από τους ε, Πράσινους ε, και θα ρωτήσω την Σαμπίνη τον Πασκάλ ποιος θα πάρει το λόγο για το ΕΛΚ. Θε κάτι να προσθέσει. Ναι, θέλω να ζητήσω συγγνώμη που πρέπει και εγώ να αποχωρήσω. Δεν πάω στην τουαλέτα. Έχω ε, μία συνάντηση με την Προεδρία για ένα σημαντικό θέμα. Ζητώ συγγνώμη. Θα δώσω το λόγο και παρακαλώ όλους σας να είσαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. για να δώσουμε χρόνο στον Επίτροπο να απαντήσει. Καθυστερούμε, αλλά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μέχρι τις 12 και 10, το τελευταίο 20 λεπτό. Θα ήθελα να το κρατήσουμε για να συζητήσουμε την έγκριση τύπου για τα οχήματα, διότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για τους ε, καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τζούλια και η Σαμπίνη Πασκάλ, ποιος θα πάρει το, το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλώς ορίσατε. Ε, εγώ θα μείνω να ακούσω την απάντησή σας πρώτα-πρώτα. Συμφωνώ με όσα είπατε για την φορητότητα, τον Μην Είναι σημαντικό να είμαστε πρωτοπόροι. Το Μάιο ευτυχώ θα έχουμε κάποιες προτάσεις για γεωποκλεισμό ηλεκτρονικό εμπόριο και φάνηκε από την διαβούλευση ότι οι καταναλωτές αυτό που θέλουν είναι τον αποκλεισμό ε, σε σχέση με το περιεχόμενο. Ξέρουμε ότι το copyright τώρα πήγε για Σεπτέμβριο και αυτό δεν αλλάζει. Όμως πρέπει να σας πω ότι η οδηγία για καλωδιακή και δορυφορική θα μπορούσε να ε, έχει τύχει διεκπαιρέωση νωρίτερα. Τώρα, ε, άσχετα δηλαδή από τη δέσμη copyright, τα είπαμε για τη συνθήκη του Μαρακές, έχουμε και κάποια στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα, γιατί μπήκε στο ψυγείο για το τελευταίο τρίμηνο η συνθήκη. Αλλά αν κατάλαβα καλά, εσείς θα την διεκπαιρεώσετε τον Σεπτέμβριο μαζί με τη δέσμη για το copyright. Βέβαια θα πρέπει να είναι διαφορετική δέσμη μέτρων γιατί για τη συνθήκη δεν υπάρχει καμία προστριβή. Ε, και ελπίζουμε ότι τελικά θα εφαρμοστεί με κανονισμό για μην αργήσει άλλη μια διετία η υλοποίηση και εφαρμογή της. Τώρα για το copyright έχουμε την πρόταση, έχουμε την πρόταση για ε, καλώδιο και δορυφόρο, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμόσει την οδηγία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οδηγία, με άλλο τρόπο. Α, μας είπατε για την εκπαίδευση και τις βιβλιοθήκες. Αλλά τι γίνεται με την έρευνα. Γιατί για την έρευνα υπάρχει θέμα όσον αφορά τους ερευνητές. Άρα, για πέστε μας, θέλετε μια γενική εξαίρεση που τα καλύπτει όλα αυτά ή πολλές επιμέρους εξαιρέσεις. Είπε ο συνάδελφος ε, Ντάλτον επίσης ε, την πιθανότητα τέλους για το YouTube. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω δεν θέλετε να αναθεωρήσετε την ε, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ανέβασμα στο ίντερνετ κάποιων βίντεο ε, που δεν επιδέχονται τέλος. Δεν ξέρω. Διευκρινίστε μας. Τι θα γίνει με τον ασφαλή λιμένα, με τη σχετική αρχή. Θα ισχύσει. Επίσης μας εξέπληξε η απόφαση της Επιτροπής να κάνει την διαβούλευση για επικουρικά θέματα copyright. Εμείς έχουμε καταψηφίσει από ένα χρόνο με αφορμή την δική μου έκθεση τέτοιε κινήσει. Άρα τώρα ζητάει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκδότε για δημοσίευση των τύπων αλλά και για πάσα δημοσίευση. Εμεί είχαμε πει όχι σε αυτό. Και τώρα Ίσως γι' αυτό πάγωσε η πρόταση για το copyright. Είπε βέβαια ότι είναι η ύψιστη προτεραιότητα για την τρέχουσα επιτροπή ο πρόεδρος Γιούνκερ. Πρόεδρος. Σαμίν. Ναι, και από δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Επίτροπο για την ανταλλαγή αυτή απόψεων εκ νέου. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια ζητήματα. Καταρχάς, την φορητότητα. Πολλές φορές ακούσαμε ήδη ότι κυρίως η επαλήτευση του συνήθους τόπου διαμονής αποτελεί σημείο κλειδί στο θέμα αυτό. Ε, τι πιστεύετε σε ό,τι αφορά το χρονικό όριο ότι δεν έχει νόημα, ναι, αλλά υπό τον όρο ότι ο συνήθις τρόπος, τόπος διαμονής του συνδρομητή θα είναι σαφής. για να ρυθμιστούν και τα θέματα της δεσμευριακής πρόσβασης. Είπατε επίσης ότι σε, επί της αρχής ε, αποδέχεστε την αρχή της ε, ε, εδαφικότητας σε ό,τι αφορά τις άδειε προς τις εταιρείε σε ό,τι αφορά τον οπτικοακουστικό κλάδο. Θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τον κλάδο αυτό έχει δικαίωμα να κάνει συγκεκριμένες ε, προτάσεις προδιαγραφών και πόσο σημαντικό αυτό είναι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων που θέλουν να προσφέρουν τέτοια περιεχόμενα. Και περνάω στο δεύτερο σημείο, σε ό,τι αφορά το αδικαιολόγητο γεωποκλεισμό σε πολλούς ε, τομείς, ε, μέσω ψηφιακή κάρτα, μέσω διεύθυνση IP Αφενός λοιπόν έχουμε τα θέματα φορητότητας που, προ... που προκαλούν τέτοιες διακριτικές μεταχειρήσεις ε, σε ό,τι αφορά τον τόπο και από την άλλη τα καταργούμε αυτά. Θα πρέπει να υπάρχουν όμως σαφείς ορισμοί του πεδίου εφαρμογής στους, στα εκάστοτε νομοθετήματα και υπάρχουν ε, για παράδειγμα συγκεκριμένα α, παραδείγματα. Οι Ολλανδικοί σιδηρόδρομοι, για παράδειγμα, μπορούμε να αγοράσουμε εισιτήριο online, αλλά μόνο με Ολλανδική κάρτα, όχι με Γερμανική ή Βελγική κάρτα. Πραγματικά πολλά ακόμα είναι κρεμή και πραγματικά σας υποστηρίζουμε. Αυτό που είναι σημαντικό για την ε, στρατηγική είναι να προχωρήσει και η ανάπτυξη των υποδομών, ε, υψηλές συχνότητες, γιατί και στο σημείο αυτό μεταξύ κρατών μεταξύ κρατών υπάρχουν τεράστιες διαφορές και σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους χώρους ε, ε, στο σημείο αυτό. Πώς λοιπόν αυτές οι μεγάλες διαφορές τα επόμενα χρόνια μπορούν κάπως να αμβληθούν και τι πιστεύετε σε ό,τι αφορά και τον ανταγωνισμό στις τηλεπικοινωνίες. Στην παρούσα φάση στη Γερμανία έχουμε με τον vectoring ε, ε, το οποίο οδηγεί σε εκ νέου μονοπόλια. Τα έχει αυτά στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Από το καλοκαίρι και μετά θα μας απασχολήσει και μάλιστα πολύ. Το θέμα είναι λοιπόν ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα πέντε εφαρμογής, ποιοι εμπίπτουν σε αυτό γραμμικές υπηρεσίες θα συνεχιστούν ή όχι, τι νόημα έχει το θέμα της προστασίας των, της νεολείας το θέμα της προστασίας του καταναλωτή, των διαφημίσεων. Και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Καλά θα τα ακούσουμε και κάποιες βασικές ιδέες. Σε ό,τι αφορά το copyright, τα πνευματικά δικαιώματα, ε, εξαιρέσεις, ε, περιορισμοί, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όμως ε, Ποια είναι η άποψη τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και πώ σκοπεύετε όλα αυτά να προστατεύσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι επόμενοι μιλητέ από ένα λεπτό καθένα όμω. Ένα λεπτό ο καθένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για το όσα μα είπατε. Νομίζω ότι θα μπορούσα να ολοκληρώσω μέσα σε ένα λεπτό. Όσον αφορά τα απτά αγαθά, ε, κάποιο που αγοράζει αυτή τη στιγμή επιγραμμικά το ίδιο προϊόν με κάποιον που το αγοράζει ε, αλλού έχει περισσότερα δικαιώματα. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο ε, είναι λογικό το να έχουμε αυτή τη διάκριση. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Γιατί η Κομισιόν δίνει περισσότερα δικαιώματα σε όποιον αγοράζει επιγραμμικά και δεύτερον η Ευρωπαϊκή Επίτροπη ήδη ανέφερε ότι θα πρέπει να ε, προσαρμόσει την σχετική οδηγία στο πλαίσιο του REFIT. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα Μέχρι τότε θα έχουμε ε, ε, αναθεώρηση της οδηγίας. Επίσης, μιλήσατε για φορητότητα ε, του επιγραμμικού περιεχομένου, μιλήσατε για τους ανθρώπους που κάθε μέρα περνούν τα σύνορα για να εργαστούν αλλού. 1,7 πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνουν αυτό. Είναι αρκετά μικρό ποσοστό σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό. Είπατε ότι δεν βρίσκεται πολύ καλή η ιδέα να περιορίσουμε τον αριθμό, τον αριθμό ημερών για την φορητότητα. Και επίσης ε, αναφερθήκατε στο fair use και τον ορισμό ε, της ζωστής ε, χρήσης. Ο διευθυντής της Πρόξιμους της βελγικής εταιρείας εκείνη της τηλεφωνίας είπε ότι θα περιορίσει αυτό το fair use σε 50-60 μέρες, ε, αλλά ε, κάποιος που περνάει τα σύνορα κάποια μέρα τιμωρείται διπλά. Πρώτον, επειδή πρέπει να περάσει το σύνορα για να δουλέψει και α, από την άλλη, επειδή ουσιαστικά ε, δεν δικαιούται αυτή την κατάργηση του, της περιαγωγής. Θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο και να έχει ε, το περιορισμό αυτών των 50-60 ημερών. Ευχαριστώ, Βίκη. Κύριε Αντιπρόεδρε, πρώτα-πρώτα. Περιμένω να βάλετε τα ακουστικά. Όσον αφορά το θέμα το οποίο τώρα μας απασχολεί και εσείς έχετε ασχοληθεί, όσον αφορά το δίκαιο του καταναλωτή για τα ψηφιακά. Πολύ καλό να έχουμε ρύθμιση πάνω σε αυτό, αλλά στην πρότασή σας ε, έχετε αφήσει πολλά κενά. Συγκεκριμένα το πώς θα έχουμε συνέπεια, συνοχή μεταξύ των επιμέρους νομοθετημάτων για τα ψηφιακά και τα μη ψηφιακά, τα απτά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε κάποιες επικαλύψεις και κάποια σημεία που υπάρχουν κενά στη ρύθμιση. Συμφωνώ με την ανησυχία της Εύελιν, ότι δηλαδή αν έχουμε δύο καθεστώτα προστασίας καταναλωτή που συνεπάρχουν. Έχουμε δηλαδή μια συγκεκριμένη προστασία για τις ε, ιντερνετικές αγορές. Οπότε θα πρέπει να καταλάβει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις ο καταναλωτής. Οπότε νομίζω ότι άλλους θα εξυπηρετήσει αυτή η ρύθμιση και όχι τους καταναλωτές. Όσον αφορά τη φορητότητα είναι θέμα όντως της ε, διάρκειας αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εδαφικότητα δεν θα πειραχτεί. Γιατί με την αρχή της εδαφικότητας τώρα μπορούμε να έχουμε την συνέργεια όλων των εμπλεκομένων ε, που βοηθούν για το πολιτικό περιεχόμενο. Άρα θα πρέπει για να υπάρχει εξακρίβωση του τόπου συνήθους διαμονής. Έχουμε τον σημερινό κανονισμό, ο οποίος όμως δεν είναι ξεκάθαρο για αυτό το θέμα. Μας είπατε τώρα και για το YouTube. Ε, τα δύο τρίτα των βίντεο εκεί αντιπροσωπούν το 10% της αμοιβή των δημιουργών, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά την οικονομική διάσταση του φαινομένου YouTube. Κυρία Κάλλας. Μια σύντομη ερώτηση. Δεν σχετίζεται άμεσα με αυτά τα οποία είχατε προτείνει, αλλά έχει σχέση με την οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου. Ρωτώ, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή τη οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπορίο. Διότι είδαμε σε διαφορετικά κράτη-μέλη ότι έχει αναπτυχθεί προβληματική και Ε, υπάρχει ανομοιογενής εφαρμογή ή ορισμοί ας πούμε τι πάει να πει ε, παράνομο περιεχόμενο κλπ. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Έχω εδώ ένα κατάλογο με ερωτήσεις. Απαντήστε όπου μπορείτε για προστασία των δεδομένων Ναι, θα χρειάζονται κατευθυντήριε γραμμέ και να δούμε τι γίνεται με το ψηφιακό περιεχόμενο. Θα πρέπει να έχουμε προσέγγιση αποδοτική και να μην υπάρχει σύγκρουση των εμπλεκομένων στα ψηφιακά με, το, με τους εμπλεκόμενους στο GDPR. για την ευθύνη του ενδιαμέσου και τις πλατφόρμες υπάρχουν όντως επιμέρους ευθύνες. Θα πρέπει να μην περιπλέξουμε τα πράγματα για τους ε, ενδιάμεσους. Για την τυποποίηση και προτυποποίηση. Μιλήσαμε χτες με αφορμή το TTIP, τότε θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την επέκταση της ψηφιακής τεχνολογίας και να μην έχουμε κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία να διαφέρουν από τα αμερικανικά πρότυπα με τα διεθνή πρότυπα. Άρα, για πετε μας εσείς τι έχετε υπόψη σας. Πολύ σημαντικό αυτό. Για τον γεωαποκλεισμό δεν θα πρέπει να έχουμε δεσμενή διάκριση από την ενιαία αγορά, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει οι εταιρείε να υποχρεώνονται να έχουν ίδια τιμή σε όλα τα καταστήματα παντού στην Ευρώπη, γιατί θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν επιλογή ελεύθερη. Αυτά ήθελα εγώ να ρωτήσω γιατί τα συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να προσέξουμε με τους ε, ορισμούς για τις πλατφόρμες. Υπάρχει ποικιλία και στις πλατφόρμες ανά τομέα. Θέλετε τώρα να απαντήσετε και βεβαίω μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση με το ίντερνετ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μου φαίνεται ότι δεν χρειάζεται να δώσω απαντήσεις. Γιατί η κυρία Βίκη Φόρτ έχει συνοψίσει πραγματικά τις απαντήσεις μου και τις σκέψεις μου. Δεν ξέρω τι κάνω σε αυτή τη συνεδρίαση. Περιτεύω. Έχουμε ακριβώς τις ίδιες απόψεις όπως και να έχει. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω, αλλά να μου πείτε πότε θα πρέπει να ολοκληρώσω τα καταληκτικά μου σχόλια. Σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες, γιατί ξεκινάω από, την... το σημείο αυτό. Έχετε δίκιο, γιατί λέτε ότι έχουμε διαφόρων ειδών πλατφόρμες και ο κόσμος, ε, όταν μιλάει για πλατφόρμες, είναι διαφορετικά πράγματα. Κάποιοι, για παράδειγμα, έχουν υπόψη ε, μηχανές αναζήτησης. Ε, και εδώ θέλουν διαφάνεια. Θέλουν να ξέρουν ε, ποιες μηχανές αναζήτησης προωθούν ποια προϊόντα. Και πού μπορεί κανείς να βρει πραγματικά τους, τις κορυφές τη της αγοράς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε κάποιες ε, πληροφορίες παραπάνω σε αυτά τα άτομα που ζητούν διαφάνεια. Κάποιοι άλλοι όταν μιλάνε για πλατφόρμες μιλάνε κυρίως για θέματα προστασίας καταναλωτή κυρίως για παράδειγμα τους ταξιτζίδες. Και φυσικά όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να σεβόνται τους κανόνες μας. Αλλά εμείς ε, ως πολιτικοί θύνοντες θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η οικονομία θα μείνει, γιατί υπάρχουν νέες τεχνολογίες και οι νομοθέτες θα πρέπει και αυτοί να προσαρμοστούν. Είναι απόλυτα απαραίτητο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε οποιαδήποτε σχέδιο να καταπνίξουμε την καινοτομία και να ρυθμίσουμε τις πλατφόρμες αυτές. Άρα, κάποιοι άλλοι όταν λένε πλατφόρμες, βασικά σκέφτονται ε, πλατφόρμες που για παράδειγμα παρέχουν μουσική μέσω συνδρομής. Τέτοιες ε, πλατφόρμες ε, ε, αποφέρουν ε, 1,6 δισεκατομμύρια στους ε, παραγωγούς, στους δημιουργούς, όπως το Spotify. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες που υποστηρίζονται από διαφημίσεις, όπου υπάρχουν ένα δις επαφές ανά μήνα. Αλλά αυτές οι πλατφόρμες ε, αποφέρουν πάρα πολύ λίγα μόνο 0,6 για παράδειγμα στους δημιουργούς. Φυσικά, πλατφόρμες αυτές ε, λένε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται στις πλατφόρμες μας. Εμείς τίποτα, ουδέτεροι διαμεσολαβητές είμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει λίγο παραπάνω σαφήνεια. Πού μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά κάποιος είναι ουδέτερος διαμεσολαβητής και πού ε, πρέπει να πούμε, κοιτάξτε, όχι, ε, Πωλείτε πραγματικά προϊόντα χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο κάποιου δημιουργού χωρίς να τον ε, πληρώνετε. Δεν κατηγορώ οποιαδήποτε πλατφόρμα, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο σαφείς κανόνες. Γιατί όταν τα πράγματα είναι άσπρα και η μαύρα, είναι σαφές τι γίνεται. Αν υπάρχει παράνομο περιεχόμενο, για παράδειγμα. Αλλά αν το περιεχόμενο είναι νομιμό, αλλά σε κάποιες πλατφόρμες ε, χρησιμοποιείται με παράνομο τρόπο, ε, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και είναι δύσκολο και παίρνει χρόνο μέχρι να κατέβει για παράδειγμα το τραγούδι από το ίντερνετ. Και είναι πολύ άμεσα η ανταπόκριση του κόσμου που το βάζει, για παράδειγμα, σε μια άλλη πλατφόρμα. Θα πρέπει να ακούμε τι λένε και οι μουσικοί που διαμαρτύρονται. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα της αμοιβή, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό φυσικά. Αλλά το θέμα είναι πώς θα έχουμε και ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ε, ιστοσελίδων των πλατφόρμων εκείνων που ε, χρησιμοποιούν διαφημίσεις και αυτών που χρησιμοποιούν ε, σύνδρομες. Άρα προσπαθήσαμε να μην ακολουθήσουμε οριζόντια προσέγγιση, να μην προσπαθήσουμε να τα ρυθμίσουμε όλα, όλες τις πλατφόρμες με ένα κανονισμό. Είναι αδύνατον. Σε ό,τι αφορά τον ασφαλή λιμένα θα παραμείνει ως έχει αποφασίσαμε να εξετάσουμε τα προβλήματα ένα προς ένα. Κατά περίπτωση να βρούμε λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα. Όχι να αλλάξουμε εκβάθρον τις ε, βασικές αρχές του διαδικτύου. Για τον γεωποκλεισμό τώρα. Η πρόταση αυτή το sell like at home, το πωλήσει δηλαδή όπω και στην ημεταπή, δεν έχει να κάνει με τι ίδιε τιμέ παντού. Έχει να κάνει με την ελευθερία του παρόχου, του πολιτή. όπω ξέρετε και στα καταστήματα οι τιμέ μπορεί να είναι διαφορετικέ. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Και αυτό θα παραμείνει έτσι. Θα υπάρχει ακόμα διαφοροποίηση στι τιμέ, αλλά οι καταναλωτέ θα πρέπει να μπορούν να έχουν την ε, επιλογή. Αν κάποιο ζητά υπερβολικά υψηλή τιμή, εγώ ως καταναλωτή θα πρέπει να έχω δικαίωμα να πάω σε άλλο online κατάστημα, σε άλλη ιστοσελίδα. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει ως δυνατότητα και πάλι θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η υποχρέωση της πώληση όπως την ημεδαπίδα θα πρέπει να είναι υποχρέωση και παράδοση των προϊόντων. Θεωρώ ότι αυτό τι θα σημαίνει ότι θα υπάρχει αυτή η αρχή σε ό,τι αφορά τις πωλήσει. Τώρα αυτό που θα συνδέεται με την Ρώμη 1. Το είχαμε ξεκαθαρίσει, αλλά η λύση αυτή θα είναι απλή και ξεκαθαρή. Οι πολιτές ε, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις ε, ετικέτες αυτές της επισήμωση αυτή. αν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, θα μπορώ να επιστρέψω, για παράδειγμα, τις συσκευές που αγόρασα στην, ε, στο μέρος που τις ε, αγόρασα. Και ο πολιτής δεν χρειάζεται να ανησυχεί το πώς θα συγκεντρώσει τις συσκευές από τις τέσσερις γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ιδέα που αναπτύσσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα τυποποίησης, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ε, ανοιχτά πρότυπα στους διάφορους τομείς. Πριν από δύο μέρες συναντήθηκα με τον Τζένι Ρομέτσι από την IBM. Η IBM είναι σχεδόν ευρωπαϊκή εταιρεία. Γιατί? Πάνω από 100 χρόνια δραστηριοποιούνται εδώ και γνωρίζουν εις βάθος την ευρωπαϊκή αγορά και κατανοούν ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη να δημιουργηθεί μαζί με τους Αμερικανούς ένα πλαίσιο ανοιχτών προτύπων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν για το διαδικτύο και πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε πάνω από 600 διαφορετικά πρότυπα που καλύπτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ζητήματα αυτά. Για τις μικρές επιχειρήσεις είναι αδύνατον, εντελώς αδύνατον να κατανοήσουν όλα αυτά τα πρότυπα. Και σύμφωνα με όσους ε, παράγουν ε, και συσκευέ. για παράδειγμα, αυτό τι δείχνει, ότι αν θέλουμε να συνδέσουμε το ψυγείο με την σκούπα την ηλεκτρική και το πλήρω πιάτων, θα πρέπει να μπει ένα τσιπάκι μέσα στις συσκευές αυτές. Η τιμή δε για το τσιπάκι αυτό είναι 50 ευρώ. 50. διατείνονται ότι αν ε, υπάρχουν ανοιχτά τα πρότυπα, η τιμή θα είναι μόνο ένα ευρώ για τη διασύνδεση όλων αυτών των συσκευών. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι γιατί οι καταναλωτές να πληρώσουν 49 ευρώ παραπάνω Όλα αυτά καταλαβαίνετε τι σημαίνουν για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Θα θέλαμε να υπάρξει να ξεκινήσει μια διαδικασία τυποποίηση. Η τυποποίηση θα πρέπει να παραμείνει όσο έχει. Είναι μια εθελούσια διαδικασία την οποία την προαγάγει ο βιομηχανικός ο οικονομικός κλάδος. Θα πρέπει να μείνει λοιπόν έτσι. Αλλά θεωρούμε ότι σε κάποιε περιπτώσει σε, σε κάποιους τομείς προτεραιότητας μπορούμε να επιταχύνουμε τα πράγματα. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε για την ευθύνη του διαμέσου λάβετε, Το έθιξα το θέμα αυτό. Δεν θα υπάρξει οριζόντια προσέγγιση. Το safe harbor ασφαλής λιμένες θα πρέπει να παραμείνει όσο έχει αλλά θα πρέπει να είναι πιο σαφείς οι κανόνες. Δεν έχει νόημα να κατηγορούμε κάποιες ε, κακές, σε εισαγωγικά, πλατφόρμες. Και να τελικά να μην κάνουμε τίποτα. Δεν είναι σκόπιμο αυτό ως ιδέα. Και ύστερα φυσικά δεν έχουμε οποιοδήποτε πρόθεση να βάλουμε φόρο στο YouTube κτλ. Αυτό το άκουσα από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούω ότι συζητούν τέτοιους φόρους για το YouTube, αλλά πολύ απλά να σας πω ότι λυπάμαι, εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα συζητούν αυτά. Και πολύ αμφιβάλλω κατά πόσον πραγματικά συζητιούνται αυτά. Εγώ ποτέ δεν υποστήριξα ιδέες τέτοιες. Επαναλαμβάνω όμως ότι αν υπάρχει ανάγκη θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες μας, να τους κάνουμε πιο σαφείς. Φορητότητα. Όχι, δεν θα υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ανά ημέρα. Γιατί είναι περιτά. Αλλά η συνδρομή θα πρέπει να αποτελέσει τη διαχωριστική γραμμή. Η ταυτοποίηση τώρα είναι σημαντικό ασφαλώ τμήμα τη διαδικασία αυτή. Άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε το αρχή τη εδαφικότητα. Και αυτό γιατί η χρηματοδότηση νέων ταινιών βασίζεται στην αρχή της εδαφικότητας. Εγώ δεν είμαι κατά της αρχής αυτής της εδαφικότητας, αλλά είμαι κατά της αυταρχικής αποκλειστικότητας. Κάποιος κόσμος λέει και ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να παρέχουμε στους ενεχόμενους επενδυτές απόλυτη αποκλειστικότητα εδαφική όσο έχει σήμερα. Μα σήμερα, να μας συγχωράτε, δεν υπάρχει αυτή η αποκλειστικότητα η εδαφική η οποία διατείνεται ότι υπάρχει. Τι γίνεται με το 20% των χρηστών ε, διαδικτύου που χρησιμοποιούν το VPN ή 68% που χρησιμοποιούν τα δωρεάν α, συστήματα για να κατεβάζουν ταινίε. Άρα, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση απορριτή εδαφική αποκλειστικότητα και όσοι παρέχουν σε κάποιον ε, απόρριτη εδαφική αποκλειστικότητα σήμερα. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους θα ήθελα να πω ότι απλά ψεύδονται. Καταφανώς γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Σκοπός μας είναι να δώσουμε νόμιμη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Και σκοπός μας είναι να παρέχουμε και μία σωστή δίκαιη ανταμοιβή στους δημιουργούς. Νομίζω ότι δεν έχω επαρκή χρόνο για να απαντήσω για τα υπόλοιπα, αλλά ε, μόλις ξεκίνησα και χρειάζεται να μιλήσουμε και για το θέμα των αυτοκινήτων, λέει η Πρόεδρος. Το επόμενο θέμα μας, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνετε, Επίτροπε. 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι που εργάζονται σε άλλα κράτη-μέλη για το θέμα της φορητότητας, το είπαμε. Ε, και αυτό το είπαμε, τη συνεργατική οικονομία και αυτή την αναφέραμε. Η Επιτροπή αυτή δεν σκοπεύει να καταπνίξει την καινοτομία μέσω υπερβολικής ρύθμισης. Το είπα και αυτό. Τόσες ερωτήσεις, τόσες ερωτήσεις. Κάθε βουλευτής τουλάχιστον 5-15 θέματα έθιξε. Και είναι δύσκολο πραγματικά να τα απαντήσω όλα, γιατί συχνότητες τέθησε ένα ερώτημα όμω. Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες. Για το πώς ε, να προβλέψουμε το ανώτατο όριο 700 MHz, γιατί πραγματικά ένα μεγάλο τμήμα ε, του το ε, ποσοστό του τμήματο αυτού είναι αξιοσημείωτο και κάποιε χώρε ζήτησαν μια μεταβατική φάση. Αλλά κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ανταγωνισμό και όχι μόνο ανταγωνισμό εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παγκόσμιας κλίμακα ανταγωνισμό. Και βέβαια μπορούμε να τα παρέχουμε αυτά. Και φυσικά μπορούμε να προβλέψουμε μεταβατική περίοδο 2 ετών, 20 ετών άμα θέλετε. Αλλά τι θα σήμαινε αυτό, τι θα σήμαινε μία τέτοια μακρά μεταβατική περίοδος. Βρισκόμαστε πραγματικά σε μία περίοδο που πρέπει να βιαστούμε, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Βιαζόμαστε γιατί μιλάμε για το μέλλον μας. Και αν κάποιος θέλει να καθυστερήσει, θα το πληρώσουμε αυτό στο μέλλον. Αυτό εξαρτάται από τους πολιτικούς ευθύνοντες, αλλά εγώ δεν είμαι υπέρ τέτοιων ιδεών. Πρόεδρος. Α, συμπαθάτε συμπαθάτε Α, για το copyright. Δεν ξέχασα να σας πω. Ήταν σημαντικό, λέει ο Επίτροπος, γιατί ξεκινήσαμε ακόμη μία δημόσια διαβούλευση. Γιατί κάποιοι εκδότες ζήτησαν επικουρικά δικαιώματα copyright Αλλά ούτε στη Γερμανία δεν είναι ξεκαθαρή κατάσταση. Ορισμένοι λένε ότι με τίποτα δεν θέλουμε επικουρικό copyright και ανακαλύπτεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι έχουμε κάποια προβλήματα ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο να σκεφτείτε την άλλη Gemeine Zeitung Και υπάρχουν επομένω πολλέ απόψει και μέσα στην Γερμανία. Πολλοί εκδότε επομένω ζήτησαν να ασχοληθούμε με τα γειτονιάζοντα, γειτονικά δικαιώματα. Αυτά ισχύουν για τη μουσική, αλλά όχι για τους εκδότες. είπαμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο προς το παρόν. Τα έχουμε συζητήσει πάντως. Έχουμε τα στοιχεία για να λάβουμε την απόφαση. Αλλά όταν έγινε η διαβούλευση, το συγκεκριμένο θέμα δεν έφυγε. Επίσης, υπήρχε και το θέμα της ελευθερίας πανόραμα. Το λεγόμενο πανόραμα η σχετική ελευθερία δεν συζητήθηκε κατά τις διαβουλεύσεις. We discussed enough. Now... Έγινε αρκετή συζήτηση, ε, λένε και τώρα ήρθε να αποφασίσει. Άρα θα διατυπώσουμε κάποια πρόταση το Σεπτέμβριο. Άρα έτσι θα δοθεί συνέχεια σε αυτές τις διαβουλεύσεις. 200 uh, <laughs> uh, uh, ε, Είναι όλα αυτά δύσκολα, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα, λέει ο Επίτροπος. Πάντως χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Συνεχίζουμε. Είχαμε ε, πάρα πολλές ψηφοφορίες που κράτησαν πάρα πολλή ώρα, για πάρα πολλή δυσκολίες σήμερα το πρωί. Οπότε και γι' αυτό το λόγο έχουμε μείνει πίσω για το χρονοδιάγραμμα μας. Οπότε πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας με τη διάταξη. Είναι παρουσίαση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ε, έγκριση και έλεγχο της αγοράς για τα οχήματα με κινητήρα και τα ρημουλκούμενα. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρουσίαση για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ακούτε! Και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε αρκετό χρόνο για να το συντηρούμε στην Επιτροπή μας. Ευτυχώς έχετε έρθει κύριε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συχτής λέει ότι δεν θέλουμε τίποτα να το συζητήσουμε βιαστικά. Εάν θέλετε να το αναβάλουμε για άλλη συνεδρίαση, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε στις 24 Μαΐου. Σε ένα μήνα δηλαδή. Μπορείτε να αρχίσετε την εισήγησή σας ε, από πλευρά Επιτροπής. Αλλά το 20 που μας απομένει δεν αρκεί. Ξέρω επίση ότι κάποιοι ασχεδόν ηγητέ πρέπει να σπέψουν στο αεροδρόμιο. Τι λέτε. Θέλετε να αρχίσετε να διακόψουμε και να μας τα ξαναπείτε, ε, να συνεχίσουμε τέλο πάντων σε ένα μήνα. Έχουμε ως μισή ώρα. Χρειάζεται μισή ώρα και ίσως και παραπάνω για να το πούμε σωστά. Εσείς τι λέτε από την Επιτροπή. Thank you very Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνουμε τον χρονικό περιορισμό που υπάρχει, ωστόσο πιστεύουμε ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από εσάς και τον εισηγητή όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε. Πρόεδρος, ε, να προτείνω εγώ τότε η παρουσίασή σας υπάρχει στο διαδίκτυο. Μπορούν λοιπόν οι ευρωβουλευτές να αρχίσουν να τη διαβάσουν, να ξεκινήσουν τις άτυπες συζητήσεις και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση στις 24 Μαΐου. Εντάξει. Συμφωνεί και ο εισηγητής. Ε, ναι, μόνο να πω ότι ε, έχω δει την παρουσίαση αυτή. Είναι πολύ μακροσκελής και πλοκή. Δεν θα έχουμε το χρόνο να τη συζητήσουμε τώρα, ωστόσο θα ήθελα να ε, προσθέσω ότι η καθυστέρηση του ενός μήνα στην Επιτροπή δεν σημαίνει καθυστέρηση της συνολικής ε, διαδικασίας, ε, διότι ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να υποβάλουμε πρόταση πολύ σύντομα. Η κυρία Σκάλτεμοζεν, συμφωνώ, νομίζω ότι θα πρέπει να αναβάλουμε το θέμα αυτό στις 24 Μαΐου και κάτι ακόμα. Όπως ε, γνωρίζετε και ο κύριος Ντάλτον και εγώ συμμετέχουμε στην Επιτροπή ΙΜΗ, την Επιτροπή διερεύνηση του σκανδάλου τη Volkswagen. Θέλουμε λοιπόν χρόνο να δούμε τι ευρήματα, σε τι ευρήματα θα καταλήξει αυτή η Επιτροπή. Ε, συμφωνώ απολύτω με την αναβολή αυτή. Ωραία και αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους ευρωβουλευτές τη Επιτροπής μας να είναι παρόντες. Συμφωνεί και το ΕΛΚ. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους για την πολλή δουλειά που κάναμε σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ.